Έχουμε μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρίση τιμών στον ευρωπαϊκό τομέα χειρίου κρέατος. Πρόκειται για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου και καλό τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Σεκέρσκι, συντάκτη της ερώτησης, να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση ενός σοβαρού θέματος, περίπλοκου θέματος, γιατί είναι προφανές ότι ο τομέας του χείριου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει κρίση και αντίστοιχα και η παραγωγή χείριου κρέατος. Τα τελευταία χρόνια, τέσσερα χρόνια μέχρι το 2015, βλέπουμε μείωση κατά 15% των τιμών του χειρίου κρέατος. Χάρη στην ε, κοινή αγροτική πολιτική μπόρεσαν σε ένα βαθμό να σταθεροποιηθούν οι συνθήκες και ως προς το εισόδημα των ε, κτηνοτρόφων και ως προς την σταθεροποίηση της ε, προσφοράς και της ζήτησης. Ξέρουμε ότι αυτό το οφείλουμε στην κοινή γεωργική πολιτική. Και ξέρουμε ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της και ιδιαίτερα η Γεωργία της Ευρώπης ε, κρίνουν θετικά την κυνηγιορική πολιτική συνολικά. Ωστόσο η κατάσταση είναι όλο και πιο δύσκολη και τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει με τις παρεμβάσεις στην κυνηγιορική ε, πολιτική περιορίζονται ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες, την παγκόσμια δηλαδή αγορά και κυρίως την ε, παγκόσμια μείωση των τιμών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Και για να περάσω τώρα στη συγκεκριμένη ερώτηση, γνωστή σε όλους, το συνεχιζόμενο ρωσικό εμπάργκο σε εισαγωγές τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποστερεί από τον χείρο παραγωγό της Ευρώπης τη μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του. Αυτό σημαίνει σημαντικές πιέσεις μειωτικές των τιμών οι οποίες τιμές έπεσαν ε, σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που θα μπορούσαμε να δούμε σε μια περίοδο κρίσης απλώς και συνεχίζουν οι πτώσεις. Το Δεκέμβριο του 2015 είδαμε μια μείωση 9% των τιμών σφαγίων χείρων και μάλιστα στην περίοδο μέσω πριν τα Χριστούγεννα όπου συνήθως ε, αυξάνονται οι τιμές. Οι παραγωγοί λοιπόν αναγκάζονται να πολλούν και κάτω του κόστους ακόμη. Τώρα υπάρχουν τα, ε, υπάρχει η ανάληψη του τελευταίου ε, συστήματος ιδιωτικής αποθήκευσης σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, τώρα έχει κλείσει αυτό το σύστημα και δεν φαίνεται να έχει μπορέσει να σταθεροποιήσει τις τιμές. Το σερευμένο προϊόν, σερευμένο σε αποθήκες προϊόν, θα πρέπει να διτεθεί στην αγορά και έτσι αυξάνοντας την, την προσφορά θα πιέσει ακόμη περισσότερο προς τα κάτω τιμές. Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία και τι ακριβώς προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το σύστημα ιδιωτικής αποθήκευσης ε, και τις νέπιες του για τις τιμές ε, του τομέα των χοιρινών. στην Ευρώπη. Έχει αναλάβει κάποια μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να ε, ωφεληθούν οι ίδιοι οι εκτροφείς χείρων από την ε, απόδοση του συστήματος ιδιωτικής αποθήκευσης. Ξέρουμε επίσης ότι στην αλυσίδα από το αγρόκτημα στο πιάτο ε, ο γεωργός, ο εκτροφέας, ο κτηνοτρόφος είναι ο πιο δύναμος κρίκος. Πάντοτε υφίσταται τις περισσότερες συνέπειες και λιγότερο τα ωφέλη. Ξέρουμε βεβαίως ότι η απαγόρευση έχει πολιτικό περιεχόμενο σχετική με το εμπάργο το ρωσικό αλλά από την άλλη συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές για τον ε, Γεωργό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάν έχει το λόγο ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο ευρωπαϊκός τομέας χείριου κρέατος στο Όντι βρίσκεται σε μια πολύ τεταμένη κατάσταση λόγω και της ε, διεύρυνσης της παραγωγής τα τελευταία χρόνια και της απώλειας της ρωσικής αγοράς που όμως δεν είναι μόνοι λόγοι για τα προβλήματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, υποστηρίξει την αγορά με, την, με τις ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθήκευση χειρίου κρέατος. 90.000 τόνοι χειρίου κρέατος καλύφθηκαν ε, έχουν καλυφθεί με έναν προπολογισμό της τάξης των 27,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Βραχυπρόθεσμα προσπαθούμε να ε, συγκρατήσουμε την προσφορά του χειρίου κρέατος σε σχέση με τις εποχιακές τιμές στην ε, περίοδο της άνοιξης για να διοχετεύσουμε και πάλι όταν είναι πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Τώρα γιατί μπορεί να κάνει παρεμβάσει μόνο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν είναι τόσο μεγάλες ε, οι ποσότητες ε, σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά από την ιδιωτική αποθήκευση των, ε, του χειρίου κρέατος. Μπόρεσε να συγκρατήσει η ιδιωτική αποθήκευση τις τιμές και άρα τις συνέπειες στο εισόδημα του κτηνοτρόφου της Ευρώπης. Άρα αυτό το δίκτυο ασφαλείας φαίνεται να έχει φέρει αποτελέσματα και γι' αυτό θέλω ξεκάθαρα να πω ότι μέτρα της κοινή οργάνωσης αγοράς όπως η ιδιωτική αποθήκευση μπορούν αλλά δεν μπορούν, ε, ούτε μπορούν ούτε και πρέπει να αντικαθιστούν την κοινή οργάνωση αγοράς, μόνο να την υποστηρίζουν μπορούν. Και βλέπουμε σαφή ε, δείγματα ότι αντιδρά, η αγορά αντιδρά προς την ορθή κατεύθυνση. Πέραν των μέτρων στήριξης της αγοράς, ο τομέας του χείριου κρέατος έχει ωφεληθεί και από το σύμφωνο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 που προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την κτηνοτροφία εν όλο σε ύψος 400 εκατομμυρίων, 420 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα πάρα προϊόντα όπως λαρδί, λίπος και τα λοιπά και την πρόσβασή τους στην αγορά της Ρωσίας ε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε τις επίσημες αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με επιβεβαίωση και της ευρωπαϊκής ε, θέσεως και της διαπραγματευτικής θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ε, ε, πρόσβαση στην αγορά. Πιστεύουμε ότι αυτές θα ενισχύσουν δηλαδή τις θέσεις μας. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να πω ότι παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση αυτή και εάν χρειαστεί θα αναλάβουμε πρόσθετα μέτρα ταχύτατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Και τώρα από τις πολιτικές ομάδες ομιλητές με πρώτον εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του κύριο Μπούντα, Ντανιέλ Μπούντα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία ζει δύσκολες εποχές λόγω του εμπάργου προς τη Ρωσία. Ο τομέας του χειρίου κρέατος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Η παραγωγή ενός κιλού κρέατος ε, κοστίζει 1,25 και πωλείται 0,78. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Το θέμα λοιπόν είναι για ποιον δουλεύουν αυτοί οι ε, κτηνοτρόφοι. Όχι βέβαια για τις ανάγκες των καταναλωτών. Το πρόγραμμα η ιδιωτική αποθήκευση δεν είναι επαρκές για την σταθεροποίηση των τιμών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Άλλωστε σε ορισμένες χώρες τα μέτρα αυτά δεν δούλεψαν καλά όπως στη Ρουμανία. Μιας και δεν υπάρχει χώρος για την αποθήκευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βρει νέους μηχανισμούς βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά τα οποία θα στραφούν στον τομέα αυτό πρέπει να είναι ε, μεγαλύτερα από ό,τι τώρα. Επίσης, εδώ και 8 χρόνια ε, το χείριο κρέας της Ρουμανίας δεν έχει πρόβλημα σε σχέση με ζωονόσους όπως το παρελθόν και γι' αυτό θα πρέπει να μπορεί να πωλείται ελεύθερα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαράδεκτο που οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαν χρόνο για να προχωρήσουν στην εξέταση του θέματος τώρα για τους σοσιαλιστές ο κύριος Ανδρεού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε μας λέτε ότι τα εισοδήματα των ε, εκτροφέων έχουν σταθεροποιηθεί. Ζούμε σε άλλο πλανήτη. Σε μια χώρα σαν τη Γαλλία ένας γεωργός αυτοκτονεί κάθε δύο μέρες εδώ και δέκα χρόνια. Η γεωργία ζει μια βαθιά κρίση και δεν είναι γαλλικό το πρόβλημα μόνο. Παντού στην Ευρώπη χειροτερεύει η κατάσταση και αυτό που ισχύει για το χοιρινό κρέας ισχύει και για το γάλα και για τα οποροκυπευτικά. Κρίμα που δεν είχαμε μια ολομέλεια στην αρχή της εβδομάδας για την κοινή αγροτική πολιτική, για να είναι πολλοί οι συνάδελφοι και να είναι παρόν και ο κύριος Χόγκαν. Ο κύριος Χόγκαν με την απουσία του σήμερα δείχνει την περιφρόνησή του για το Κοινοβούλιο και για τους παραγωγούς χειρίου κρέατος. Το 30% των παραγωγών ζουν μια τρομερή κρίση και 10% έχουν πτωχεύσει τον τελευταίο καιρό ο κύριος Χόγκαν κάνει συστηματικά λάθος τις προβλέψεις του εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχει μια τεράστια κρίση στην αγορά και όπως ξέρετε μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρυθμιστικά καθήκοντα εδώ. Ακούστε μας πριν από το Συμβούλιο της 14ης Μαρτίου. Χρησιμοποιήστε τα άρθρα 2.21 και 2.22 για την κοινή οργάνωση που μας επιτρέπουν να πάρουμε έκτακτα μέτρα μείωσης ε, ε, παραγωγής. 3 κιλό λιγότερο ανά νεκρό ζώο θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της υπερπαραγωγής. Να ξεκινήσει εκ νέου το σύστημα ιδιωτικής αποθήκευσης ε, με έναν καλύτερο κατάλογο των προϊόντων προς εξαγωγή. Δημιουργήστε μια σωστή σήμανση ε, για το επεξεργασμένο χείριο κρέας όπως το ζητάει ο καταναλωτής και εμείς εδώ και δύο χρόνια και τέλος, ξεκινήστε μια σαφέστατη ε, διπλωματική δράση έτσι ώστε να τελειώνουμε με το εμπάργο απέναντι στους Ρώσους. Βλέπουμε ότι δεν είναι η κατάσταση εύκολη. Το θέμα δεν είναι να αναζητούμε νέες αγορές σε άλλες υπήρου, αλλά να λύσουμε το πρόβλημα με τη Ρωσία βασικά. Ευχαριστώ τον κύριο Άντρε. Για το ECR ο κύριος Βοητσεσόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των κτηνοτρόφων και των χειροτρόφων είναι πάρα πολύ δύσκολη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω όμω σε ορισμένες χώρες όπως τη χώρα μου, την Πολωνία, διότι οι χειροτρόφοι μα ε, επλήγησαν από τρία προβλήματα την πανόλη των χείρων, το ρωσικό εμπάργκο και την ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας που δεν προστατεύει τους ε, μικρούς ε, χειροτρόφους αυτούς, δηλαδή που έχουν ε, μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Η πολιτική που ακολουθείται ευνοεί τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, τα μεγάλα χειροτροφία. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Στην Πολωνία είχαμε 90 εκατομμύρια κεφαλές ε, πριν από 8 χρόνια, τώρα ούτε, τους μισού, ούτε τα μισά δεν έχουμε και πρέπει να βοηθήσουμε, ίσως να δώσουμε ενισχύσεις για ιδιωτική αποθήκευση, να βοηθήσουμε να ανοίξουν νέες αγορές ε, για το ευρωπαϊκό κρέας, Όσο πρέπει να ενισχύσουμε με επιδοτήσεις, ε, γιατί είναι μέτρα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την σήμερα δραματική κατάσταση. Οι χειροτρόφοι μας εκλυπαρούν, μας ζητούν βοήθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εκ μέρου ε, της ομάδας Άλντε, Γιάν Χοίτεμα. Για να, να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση ε, με το χείριο κρέας ε, οφείλεται και στη μείωση παραγωγής και στο ρωσικό εμπάργκο. Υπάρχει το πρόβλημα τη Αφρικανική Πανούλη των Χείρων, βέβαια. Δεν είναι νομικό το ζήτημα. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ αγορέ. Και έχουμε ακούσει και κάποια καλά παραδείγματα. Όμω πιστεύω ότι το βασικό είναι να βρεθεί μια διαρθρωτική λύση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση των ε, χειροτρόφων στην όλη αλυσίδα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να επενδύσουν ε, γιατί πρέπει να ανταποκριθούν σε υψηλότερα πρότυπα υγιεινής ε, και καλής μεταχείρισης των ζώων. Χρειάζονται επενδύσεις στις αγορές. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται σε ορισμένες χώρες ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για αύξηση της ε, παραγωγής χείρου κρέατος παρότι υπάρχει ήδη πλεόνασμα, υπάρχει υπερβολική παραγωγή και είναι πραγματικά Απορία άξιων το ότι λαμβάνεται από τον κλάδο, λαμβάνονται μέτρα ε, που δεν είναι τόσο αποδοτικά. Θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η καινοτομία. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Εκ μέρους ομάδας GUNGL, ο κύριος Μιγγέλ Φιέγας, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, Όποιο περί ανέμου θερίζει θύελε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την αγορά να ρυθμίσει όλα τα προβλήματα. Βλέπουμε τι γίνεται μετά. Χρειάζονται κρατικά μέτρα. Το 1993 η Πορτογαλία ήταν αυτάρκης και σήμερα το 40% το εσάγουμε. Οι τιμέ είναι πάρα πολύ χαμηλέ και απειλούν τον κλάδο συνολικά. Κύριε Επίτροπε, είναι επίγουσα η κατάσταση. Δεν μπορούμε με μικρά ε, μέτρα ε, διακοσμητικού χαρακτήρα να λύσουμε το πρόβλημα. Θέλουμε πραγματικά δραστικά μέτρα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη αμοιβή για τους ε, χειροτρόφους και να διατηρήσουμε το δικαίωμα κάθε χώρα να μπορεί να παράγει για να εγγυάται τουλάχιστον ε, την επισητιστική κυριαρχία. Μην επιτρέψουμε να εξαφανιστεί ένας ακόμη ζωτικός κλάδος της οικονομίας όπως τόσοι ε, χάθηκαν σε εμά τουλάχιστον μετά την ένταξή μας στην Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος εκ μέρους τώρα των Πρασίνων. Ο κύριος Ροπέ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε πίτροπε. Δεν ναι, είναι μυστικό ότι βρίσκεται σε βαθιά κρίση ο τομέας ε, του χειροκρέατος, όπως και ο γαλακτοκομικός και άλλοι. Οι τιμές ε, είναι οι χαμηλότερες ε, της δεκαετίας και η πτώση είναι 13% το χρόνο. Βέβαια οι τιμές λιανικής δεν μειώνονται. Πολλοί χειροτρόφοι πήραν ε, κάποια χρήματα για τον εξεχρονισμό της παραγωγής, για να εξασφαλίσουν ε, την ε, καλή μεταχείριση των ζώων, για να τηρήσουν κάποιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να φροντίσουμε μόνο για τη βιωσιμότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, Πού οφείλονται όλα αυτά τα προβλήματα. Πρώτον, στο ότι έχουμε μεγάλη προσφορά ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και δεύτερον, τα μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων είναι πολύ δαπανηρά. Η συμπεριφορά των εμπόρων επίσης δεν είναι πάντοτε δίκαιη. Είχαμε και την επιδημία της επάνωλης των χείρων, την Αφρικανική. Ε, άρα, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να επιδιώξουμε να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί να εφαρμόζουν οι δικοί μας κτηνοτρόφοι πρότυπα καλής μεταχείρισης και να εισάγουμε φθηνότερο κρέας, φθηνότερο κατά 25% από χώρες όπως είπα η Βραζιλία που δεν εφαρμόζουν αυτά τα πρότυπα για να μην πω ότι δεν έχουν καν αντίστοιχα πρότυπα και να μην πω τι ζωοτροφές καταναλώνουν αυτά τα ζώα από τη Βραζιλία της είπα με, ε, με μεταλλαγμένα ε, ε, Εισάγουμε λοιπόν κρέας από χώρες που έχουν ε, χαμηλότερα πρότυπα από ό,τι εμείς εδώ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πραγματική δράση. Και αυτά τα πρότυπα της καλής μεταχείρισης να τα επιβάλλει σε επίπεδο ΠΟΕ. Για όλους να ισχύουν. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ισότιμη κατανομή της προσθέμενης αξίας να περιοριστούν οι αθέμητες συμπεριφορές από εμπόρους και να μην χειραγωγούνται οι τιμές λιανικής. Επίσης να σας πω ότι σίγουρα χρειάζονται και μέτρα ενίσχυσης των εξαγωγών και ένα πρόγραμμα εγγύησης των εξαγωγών. Τέλος, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η, η νόσος αυτή που είναι πολύ εξαπλωμένη σε πολλές χώρες και ιδίως στην Λιθουανία, τη χώρα μου, έχει αποδεκατήσει το ζωικό κεφάλαιο, έχει μειώσει τι εξαγωγέ. Εμεί προσπαθήσαμε και ανακόψαμε ε, την επιδημία, αλλά ήταν πολύ μεγάλε οι απώλειε των ε, χειροτρόφων λόγω των αθέμητων εμπορικών ε, πρακτικών. Οι αγοραστέ χείρου κρέατο για υγιέστατα ζώα, τα οποία έχουν εκτραφεί στι ασφαλεί ζώνε, δίνουν πάρα πολύ χαμηλέ τιμέ για να τα αγοράσουν. Δέχεστε κύριε Ροπέ από τον κύριο Στέφαν Εκ. Γαλάζια κάρτα. Ναι, τη δέχεστε. Κύριε Εκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, θα ξέρετε ασφαλώς ότι είναι αδύνατον να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την τήρηση των προδιαγραφών για την ευημερία των ζώων εκτός της επικράτειάς της. Ερωτώ λοιπόν, θέλετε πράγματι τις προδιαγραφές για την προστασία των ζώων που με τόση δυσκολία εξασφαλίσαμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να την υποβαθμίσετε τόσο και μόνο για να έχετε πιο ε, ικανοποιητικές τιμές στην πώληση του χειρίου κρέατος. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Και θα ήθελα να πω, όπως είπα και στην ε, ομιλία μου, ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές είναι υψηλές και δεν πρέπει να δεχθούμε να γίνεται εισαγωγή κρέατος από ζώα τα οποία δεν έχουν εκτραφεί με τις ίδιες προδιαγραφές. Γιατί αυτό ε, συνιστά και αθέμητο ανταγωνισμό κατά των παραγωγών μας και βεβαίως αφορά οδηγεί σε απειλή της υγείας για τον καταναλωτή μας. Ευχαριστώ ο κύριος Κόμπορν. Απουσιάζει από ό,τι φαίνεται. Επόμενος. Επόμενη. Ομιλήτρια κυρία Ντομινίκ Μπίλντα. από την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο ευρωπαϊκός τομέας του χείριου κρέατος περνά μια δύσκολη κρίση διότι ξεπουλήσαμε τη γεωργία μας, είναι συνένοχη η πολιτική υπεύθυνη και της Ευρώπης και των χωρών. Το θέμα του ρωσικού εμπάργου είναι κάτι που καταστρέφει τους παραγωγούς στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Είναι επίγον να τερματιστεί η διαδικασία αυτή κάτι το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τις τιμές. Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας ζήτησης και προσφοράς. Η ευρωπαϊκή παραγωγή θα αυξηθεί 3% φέτος, 10 εκατομμύρια χοιρινά επιπλέον. Έτσι η Γάλλη παραγωγή πέφτουν θύματα των Ισπανών και Γερμανών παραγωγών που προχωρούν στο κοινωνικό ντάμπινγκ γιατί χρησιμοποιούν ξένους εργάτες που τους πληρώνουν 5 ή 6 ευρώ την ώρα ε, στην Γερμανία ή χωρίς κοινωνικά δικαιώματα όπως στην Ισπανία. Ε, το ανώτατο όριο είναι το 1,40 στη Γαλλία το κιλό, κάτι το οποίο ίσα ίσα μας επιτρέπει να επιβιώσουμε. Ε, φυσικά αυτή η ελάχιστη τιμή απέναντι στον ξένο ανταγωνισμό θεωρήθηκε απαράδεκτη από τους βιομηχάνους και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η προσπάθεια για την ποιότητα και την ευημερία των ζώων όπως και η Οδηγία 2008 για την προστασία των χείρων δημιουργεί προβλήματα στους Γάλλους παραγωγούς. Θα μας οδηγήσει στο να μην είμαστε ανταγωνιστικοί και να αγνοούμε τους κοινωνικούς ε, περιβαλλοντικούς κανόνες όπως στις υπόλοιπες χώρες. Πώς ε, ε, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι απασχολείται με το θέμα αυτό προχωρώντας την υπογραφή του TIP που θα εκθέσει τα προϊόντα μας στα δικά τους τα οποία έχουν κόστος παραγωγής κάτω από 40% και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί και στην σήμανση των προϊόντων μας. Κύριος Λίνξ. Ενάμιση λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερω για την διεξαγωγή αυτή τη κατεπίγουσα συζήτηση, δεδομένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, κατά την άποψή μου. Μια σοβαρή κρίση πλήττει πολλέ γεωργικέ και κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσει. Βέβαια το ότι μπήκε πέμπτη απόγευμα αυτή η συζήτηση μου φαίνεται ατυχέστατη επιλογή. Ο ρυθμός των χειροτρόφων ε, τα τελευταία χρόνια έχει πέσει κατά ένα τέταρτο και συνεχίζει να μειώνεται. Προβλήματα ρευστότητας, προβλήματα ύψους των εισοδημάτων αντιμετωπίζουν όλοι οι χειροτρόφοι της περιοχής μου με ένα ευρώ 30 λεπτά το κιλό του χείριου κρέατος δεν μπορούν να επιβιώσουν βέβαια. Πιστεύω το 2015 ένα πακέτο που διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα κράτη-μέλη ήταν μεν χρήσιμο αλλά όχι επαρκές. Πρέπει λοιπόν ε, να κοιτάξουμε και τις ευθύνες των εταίρων μέσα στην αγορά και την ε, πρόπτικη για εξωτερικό εμπόριο. Κάθε ευκαιρία που υπάρχει πρέπει να την αναγνωρίσουμε, να την εντοπίσουμε και να την ε, διεκδικήσουμε. Και ελπίζουμε ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Υποθέσεων τη Δευτέρα θα ληφθούν σοβαρές και καλές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ταχαμπελά για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι απαράδεκτο ότι διεξάγεται αυτή η συζήτηση χωρίς την παρουσία του αρμόδιου επιτρόπου κ. Χόγκαν. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Έχει καταρρεύσει το εισόδημα των χειροτρόφων και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, παίρνει καν το μέτρο της σοβαρότητας της κατάστασης. Γενικά στη Γεωργία, το Βέλγιο παραδείγματα έχει τεράστιο ε, πρόβλημα στο γαλακτοκομικό τομέα στο σύνολό του αλλά και στην ε, Φλάνδρα ιδιαίτερος το ε, χείριο κρέας. Η κατάσταση λοιπόν και συνεχίζω στα Ολλανδικά για το χείριο κρέας είναι τραγική. Κάθε κιλό κρέατος που φεύγει από το σφαγείο δίνει στον ε, κτηνοτρόφο λιγότερα από αυτός έχει δαπανίσει για να εκθρέψει το ζώο του. 1,5 ε, ευρώ θα χρειαζόταν για να μπορεί να επιβιώσει ο χειροτρόφος και τα ποσά αυτά δεν καλύπτουν καν τα όλο και το όλο και αυξανόμενο κόστος παραγωγής του χείρου. Με ζημία λοιπόν πολύ το κρέας του ο χειροτρόφος, κάτι το οποίο είναι παράδεκτο γενικά στην οικονομία εκτός από τον γεωργικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί απλώς να διασωθεί, να διασώσει ε, τον τομέα από τα σοβαρότερα προβλήματα, χωρίς όμως πραγματικά να μπορεί να δώσει απαντήσεις. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις εδώ και έχουμε πει ότι πρέπει ανάλογα με την τιμή του κόστους, ε, το κόστος παραγωγής δηλαδή, να ορίζονται οι τιμές της αγοράς. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής και πρέπει να γίνουν ε, μέτρα παρέμβαση περιορισμό της προσφοράς και να ε, λειτουργήσει ένα παρατηρητήριο τιμών για το χείριο κρέας, για την ε, τιμή παραγωγής, για, την, για τον αριθμό των σφαγίων, για τη λειτουργία των αγορών και των αποθεμάτων. Ε, και επίσης βεβαίως πρέπει να σπεύσουμε να εξασφαλίσουμε άρση του ρωσικού εμπάργου. Είναι σοβαρότατη η κατάσταση κύριε Επίτροπε. Πρέπει να σταματήσουμε πια να μελετούμε την υπόθεση και πρέπει να αρχίσουμε να λαμβάνουμε δράση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος μας Μπέλτερ. Ένα λεπτό αλσίβλιφτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ γιατί μιλάτε και εξαιρετικά τη γλώσσα μου, τα Ολλανδικά. Η κρίση στη... στον κλάδο του χείρου κρέατος ε... ψοβεί και καιρό. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είναι διατεθειμένος ο Επίτροπος να αναζητήσει εναλλακτικά μέτρα αντί της ιδιωτικής αποθήκευσης δηλαδή. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Είμαστε σε κρίση και ο κλάδος θεωρεί ότι η πρόορη σφαγή θα ήταν ένα πιο αποτελεσματικό μέτρο αντί της αποθήκευσης του κρέατος, διότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν οι τιμές και δεν θα στρεβλωθεί τόσο πολύ η αγορά, δεν θα υπάρξει μάλλον διατάξη της αγοράς. Και επίσης το άνοιγμα της ρωσικής αγοράς είναι σημαντικό. Πρέπει να δούμε τι ε, αξιολόγηση θα κάνει ο ΠΟΕ για την κατάσταση. Αν είναι αρνητική, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε γρήγορα δράση και όπως και ο πλήσας συνάδελφος θέλω και εγώ να τονίσω την ανάγκη να έχουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και εντός και εκτός Ευρώπης. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Σελίμοβιτς τώρα παρακαλώ. Οι συζητήσει οι οποίε έχουν γίνει δείχνουν ποια είναι τα προβλήματα τα οποία επικρατούν στην αγορά χειρίου κρέατος λόγω του εμπάργου της Ρωσίας. Αυτό δεν είναι εντελώς αληθές. Ήμασταν ε, ελάχιστα εκτεθειμένοι προς την Ρωσία ε, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε άλλωστε εναλλακτικέ αγορές. Το πρόβλημα είναι όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ε, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να παίρνουν βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως η ιδιωτική αποθήκευση. Ενώ θα πρέπει να πάρουν μέτρα διαφθρωτικού επίπεδου γιατί αλλιώς η κατάσταση θα χειροτερεύσει ιδιαίτερα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια πραγματική λύση, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του χειρίου ε, κρέατος στην Ευρώπη και να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα για την ευημερία των ζώων, για τις χώρες οι οποίες εξάγουν ε, κρέας ε, αυτού του είδους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Χάζενκαμπ. Ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Yes, sorry. Thank you, uh, chairman. voorzitter. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το χείριο κρέας ε, βιώνει μία μόνιμη κρίση εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα με την πανόλη, είχαμε πρόβλημα με τις ορμόνες, το ένα μετά το άλλο. Και αυτό γιατί η Ευρώπη θέλει να είναι ο αλαντοποιός και ο παραγωγός χειρίου κρέατος για όλο τον κόσμο. Θέλουν να επεξεργάζονται κρέατα για προστιθέμενη αξία. Συνεπώς λοιπόν πάρα πολλά ζώα περνούν από διαδικασίες και υφίστανται μεταχειρήσεις οι οποίες απαγορεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όμως οι απαγορεύσεις αυτές παραβιάζονται όπως η κοπή, η πρόορη κοπή της ουράς του ζώου. Η αποθήκευση είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα δεν δίνει αποτελέσματα δεν θα πρέπει να πιστεύουμε αυτά τα οποία ισχυρίζεται η, η βιομηχανία αυτή. Η βιομηχανία αυτή δεν είναι σε καλή κατάσταση όπως και τα ζώα τα οποία παράγει. Δεν πρέπει να τους δίδουμε χρήματα και νομίζω ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Πιερέκ. Ευχαριστώ πολύ. Και άλλα Ολλανδικά θα ακούσετε σήμερα. Είναι τελευταίο το σημείο αυτό στην Μεσχεία Διάταξη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλοί κτηνοτόφοι που ζουν, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις ζωοτροφές για τα ζώα τους και λόγω και του ρωσικού εμπάρκου που ελπίζω σύντομα να καταρριφθεί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν για τις οικογένειές τους υπάρχει λήψη ε, ισορροπίας. Οι τιμές του κόστους ανεβαίνουν και οι τιμές αγοράς ε, οι πώληση στην παιδική μας την περίπτωση μειώνονται. Υπάρχουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα, πρέπει να εφαρμόζουμε και όλα αυτά τα μέτρα. Άρα έχει ακριβήνει το κόστος για τους Ολλανδούς ε, κτηνοτρόφους οι οποίοι πρέπει να καταβάλουν ε, σημαντικό, ε, σημαντικά ποσά. Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν στη Δανία ή στη Γερμανία. Δεν είναι αυτό ισότιμο ανταγωνισμός. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό για την αποθήκευση. Αυτό όμως δεν μπορεί να καλύψει το κόστος. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να σταματήσουν, αλλά και αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν το επαγγελμά τους πρέπει να τους βοηθήσουν και να βοηθήσουν και αυτούς που θέλουν να εξυγχρονίσουν την εκμετάλλευσή τους. Κύριε Επίτροπε, ε, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε ε, και τα, τα, ε, τα κονδύλια που έχουμε για περιπτώσεις ανάγκες, αλλά και το σχέδιο δράσης που είχαμε πέρυσι για το πώς θα μπορούσε να είναι ένας πιο ισχυρός κρίκος στην, αρι... κρίκος στην αλυσίδα ή κτηνοτρόφι μας. Αυτό δεν πρέπει επίσης να το φροντίσουμε. Ο κύριος Κάρσκι τώρα. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η μακροχρόνια κρίση οδηγεί τους παραγωγούς μας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και επιβίωσης. Η ομάδα μας το 2014 ανέλαβε την πρωτοβουλία χάρη στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ταχύτατα μέτρα ε, για την προστασία του τομέα του χειρίου κρέατος της Ευρώπης από τις συνέπειες του ρωσικού εμπάργου και άλλα προβλήματα. Έχουμε υποστεί σοβαρότατες απώλειες από, τον, από την πανόλη των χείρων της Αφρικής και δεν έχουν μπορέσει η παραγωγή μας να σταθούν στα πόδια τους. Ιδιαίτερα όμως τραγική είναι η κατάσταση των Πολωνών χειροπαραγωγών και λόγω της περσινής ξηρασίας. η οποία επηρέασε βέβαια τις κτηνοτροφές και την παραγωγή γενικότερα. Πρέπει να αναλυφθούν ταχύτατα μέτρα. Για το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι μια βραχυχρόνια και μια μακροχρόνια λύση. Βραχυχρόνια, βραχυπρόθεσμη λύση θα έπρεπε να είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων μας. Έτσι ώστε να κατακτήσουμε νέες αγορές, ιδίως στην Κίνα. Μπορούμε να κατακτήσουμε την κινησική αγορά. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν μία άπαξ επιδότηση για τους χειροτρόφους και ο κύριος Χόγκαν θα πρέπει να γυρίσει με το αεροπλάνο όλο τον πλανήτη για να προσπαθήσει να λύσει αυτή την κατάσταση. Mm. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να βρεθούμε και μία βραχυ... μακροπρόθεσμη λύση. Γιατί ε, πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή και η ρωσική αγορά. Θα πρέπει να σας πω ότι στην Κροατία κάναμε μια ε, μεγάλη έρευνα για να δούμε αν υπάρχουν ακόμα κρούσματα τη πανόλη των χείρων και θα έπρεπε η Κομισιόν να διοργανώσει γενικά μια τέτοια έρευνα κατά την αποψή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Στέφαν Εκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο χείριο κρέας από όσο μπορεί να απορροφήσει η αγορά για διάφορου λόγου και λόγω του ρωσικού εμπάργου ε, και γιατί περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν την κατανάλωση του κυρίου κρέατος, το οποίο μπορεί να είναι πιο φθηνό, αλλά προξενεί πολλές ασθένειες. Γι' αυτό λοιπόν είναι αδύνατον να λύσουμε τα προβλήματα βράχη πρόθεσμα με την ε, διάθεση του κρέατος στο εξωτερικό. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στον ε, τομέα του γάλακτος, δηλαδή τα προβλήματα με τα οποία αντιμετωπίζουμε αποτελούν την απήχηση μιας εσφαλμένης επιλογής πολιτικής, της γεωργικής πολιτικής, παραγωγή υψηλότερη από αυτή την οποία μπορούν να αντέξουν οι αγορές. Πρέπει λοιπόν η παραγωγή να προσανατελωστεί στις ανάγκες της αγοράς και η παραγωγή χειρίου κρέατος πρέπει τέλους να αντιληφθούν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση κρέατος και θα είναι όλο και περισσότερη η χορτοφάγη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Σαντέχα ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μήνες τώρα οι γεωργοί πολλούν τα προϊόντα τους με ζημία. 15 με 20% των ε, εκμεταλλεύσεων ε, χειροτροφία στη Γαλλία βρίσκονται στα όρια της καταστροφής και βέβαια αυτό ε, ξεπερνάει τη συγκυρία του ρωσικού εμπάργου. Τι κάνει η Επιτροπή λοιπόν για να βοηθήσει τους παραγωγούς, μας, μας ώστε να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον το κόστος αυτών των διπλωματικών επιλογών. Δεύτερο διαρθρωτικό πρόβλημα είναι η ανισορροπία στην αλυσίδα των αξιών. Πρέπει το δίκαιο του ανταγωνισμού μας, να το προσαρμόσουμε για να μπορούν να ενώνουν τις δυνόμεις τους η παραγωγή μας και να πιέζουν περισσότερο ως προς τον προσδιορισμό των τιμών. Επίσης και πέραν του χείριου κρέατος, ολόκληρη η γεωργική παραγωγή διέρχεται κρίση. Για να παραμείνει λοιπόν μακροπρόθεσμα μια ισχυρή ε, γεωργική δύναμη η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση ταχύτατα. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. First, ε, και τώρα, ο κύριος Σον παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Την Δευτέρα το βράδυ μου παρόν στη συνεδρίαση με τον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα Γεωργίας, κύριο Χόγκαν. δεν υπάρχει αμφιβολία βεβαίως ότι υπάρχει σοβαρή κρίση και ότι χρειάζονται σοβαρότατες λύσεις. Έχω λοιπόν τρεις ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Χαν. Πρώτον, τον παρακαλώ να μου απαντήσει εάν ο γεωργικός τομέας, γιατί μιλούσαμε για το χείριο, αλλά γενικότερα ο γεωργικός τομέας είναι σε θέση να ανθέξει τις πιέσεις του, του ρωσικού εμπάργου. Και δεύτερον, βράχει μέσο και μάκρο πρόθεσμα. Τι προβλέψει έχετε για την αύξηση του μεριδίου αγοράς εκτός Ευρώπης Τρίτον, τι προσπάθειες έχετε αναπτύξει για την ανάπτυξη των πωλήσεων εντός της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής, ιδιαίτερος με βάση τα όσα είπαν και οι προραλήσαντες και ο προραλήσας συνάδελφος, δεδομένου ότι υπάρχει τάση να εγκαταλείπουν οι άνθρωποι την καταναλώση του κρέατος λόγω διάφορων και παράξενων και άλλων αποτελεσμάτων ερευνών που καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαμίκινς. Ο κ. Μαμίκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Επίτροπο. Στα πλαίσια της κρίσης αυτής μπορούμε να αναζητήσουμε κάποιες εξηγήσει όπως το ρωσικό εμπάργκο. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, πριν φτάσουμε στο θέμα των κυρώσεων, υπήρχε πάντα μία κρίση στον τομέα αυτό. και η χώρα μου η Λετωνία είναι αυτή η οποία υποφέρει περισσότερο από την κρίση με την Ρωσία. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε. Μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να κατακτήσουμε εκ νέου τη ρωσική αγορά. Είναι παραδοσιακή αγορά για τη Λετωνία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι για τη Λευκορωσία δεν υπάρχουν πια ακυρώσεις και δεν υπάρχει εμπάργκο. Οπότε θα μπορούσαμε να μπούμε και σε αυτήν την αγορά. Βέβαια αυτό δεν θα γίνει μέσα σε μια μέρα. Θα απαιτηθεί πάρα πολύς χρόνος. Να σας πω ότι το λετονικό ε, χείριο κρέας ήταν περίφημο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό κάποτε θα το θυμούνται μόνο τα βιβλία της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Πολωνών χειροτρόφων θα ήθελα να εκφράσω την αυξανόμενη ησυχία τους για την αποσταθεροποίηση της αγοράς του χείρου ε, στην Πολωνία και την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης και αποτελεσματικών μέτρων ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μου υφίσταται τις ε, δυνότερες συνέπειες από τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξάπλωση της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων και αυτό έχει τεράστια αντίκτυπο στα επίπεδα των τιμών. Τα μέτρα της Κομισιόν που υποτίθεται θα βοηθούσαν τους παραγωγούς δεν τους βοηθούν, δεν είναι αποτελεσματικά. Κάθε μέρα έχουν ζημία, μειώνεται ο κόστος ε, ε της ε, όλο αυξάνεται το κόστος και μειώνεται η τιμή πώληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβει μέτρα η Κομισιόν που θα έχουν πραγματικά θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση των χειροτρόφων στην Πολωνία. Μια χώρα που είναι ένα είδος ε, Ζώνε προστασία ε, για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέσα ώστε τα επίπεδα των τιμών να είναι τα πλέον ενδεδειγμένα, είπε η κυρία Γκοσεύσκα. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριο Ράντος, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αγγλουπία σε αυτό το ζήτημα, διότι πράγματι οι εκτενοτρόφοι και οι χειροτρόφοι βρίσκονται σε κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι θα γίνει ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε αυτή την αποθήκευση και να πουλάμε το καλοκαίρι το κρέας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Όμως, τα, τα κονδύλια που προορίζονται για τους κτηνοτρόφους πηγαίνουν τελικά σε αυτούς. Πρέπει η Κομισιόν να, να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ιδιωτική αποθηκεύση. Γιατί αν δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα οι κτηνοτρόφοι, είναι εκτεθειμένοι ε, στην, ε, στις μεθοδεύσεις ε, και στη χειραγώγηση από τους εμπόρους. Η παραγωγή τροφίμων είναι επίσης πολύ εκτεθειμένη και θα στηρίξω και τις υποδείξει ορισμένων ή οι οποίοι είπαν ότι θα πρέπει η Κομισιό να ε, προσπαθήσει να επιβάλλει ψηλότερα πρότυπα για τους ε, εισαγωγείς και να διευρύνει την αγορά. Η κυρία Μαρία Γκραπίνη τώρα έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση αυτή χτυπάει ε, όλη την Ευρώπη. Η πίεση στις τιμές του χείριου κρέατος οδηγεί σε μία μείωση του αριθμού των κτηνοτρόφων, των χειροτρόφων. Ε, πρέπει να δούμε το θέμα μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και στην προσφορά γιατί υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν συγκυριακά την κατάσταση. Τι κάνουμε λοιπόν στα πλαίσια της ΚΑΠ για να ξεφύγουμε από τις ευρωπαϊκές αγορές και τις γειτονικές αγορές. Εσείς κύριε Επίτροπε, δεδομένου και του χαρτοφυλακίου σας, να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο ε, για την Ρωσία Νομίζω ότι κανονικά στη θέση σας έπρεπε να είναι ο κύριος Χόγκαν και αυτό του το καταλογίζουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε μακροπρόθεσμα ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες για την παραγωγή χείριου ε, κρέατος. Τι επιτέλους θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Σκρίπεξ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε υπερηφανευόταν για την ποιότητα της εργασίας των ε, κτηνοτρόφων και χειοργών των κρατών μελών μας. Ωστόσο τώρα με την κρίση βρισκόμαστε ενώπιον του ε, ερωτήματος πώς θα δώσουμε λύσεις σε, αυτή την κρίση. Είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τους ε, γεωργούς και κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα τους χειροτρόφους. Ε, πρέπει να δώσουμε λοιπόν απαντήσεις, πρέπει να δώσουμε αποζημιώσεις και να αναζητήσουμε αγορές για να διαθέτουμε τα προϊόντα μας και σε τρίτες χώρες. Μπορεί να υπάρχουν επιδοτήσεις, πλην όμως οι χειροτρόφοι σε χώρες όπως η Σλοβακία αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. οι Σλοβάκοι Γεωργοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους παραγωγούς άλλων κρατών. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια λύση σε αυτή την τόσο σοβαρή κρίση. Ευχαριστώ Σικέρσκη πάρα πολύ στομό. Ευχαριστώ πολύ. Θα είχα κάποια σύντομα σχόλια είναι στην Πολωνία ο Επίτροπος Χόγκαν. Με πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας. Ήταν γνωστό ότι θα μετάβει στην Πολωνία σε τελευταίες έξι εβδομάδες ο κύριος Χόγκαν. Το γεγονός ότι ε, γίνεται σήμερα η συζήτηση ε, είναι φάση που έλαβε η ηγεσία του Κοινοβουλίου. Κρίμα που έγινε αυτό όμως. Αλλά ο Επίτροπος Χάν που είναι παρόν είναι και αυτός ε, ε, σε καλή θέση να, μας, ε, να μεταφέρει τις ανησυχίες των χειροτρόφων μας. Πρέπει να πούμε ότι η κατανάλωση μειώνεται στην Ευρώπη. Ακούμε συνεχώς στα μέσα μας και ενημέρωση ότι είναι κακό το κόκκινο κρέας για την υγεία μας και σίγουρα αυτό επηρεάζει πολύ την κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Υπάρχει και αυξανόμενος ανταγωνισμός ταυτόχρονα ε, από τις παγκόσμιες αγορές. Αν θέλουμε να βγούμε κερδισμένοι ε, σε αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού θα πρέπει κατά την άποψή μου να εκδομηχανίσουμε την παραγωγή. Άρα είναι δύσκολο τα μικρά χειροτροφία να παραμείνουν. Αλλά αυτό είναι ένα στόχο. Ένα άλλο στόχο είναι να παραμείνουν και να επιβιώσουν και αυτή η μικρή παραγωγή γιατί είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή αγορά. Äh, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. και ευχαριστώ πολύ για την εξήγηση γιατί ο κύριος Φαγκάν δεν μπορέσε να είναι σήμερα αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη την υπόθεση αυτή. Είναι ένα θέμα άλλωστε αυτό το χείριο Κρέατο που βρίσκεται και στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας για τη Δευτέρα. Ο κύριο Χόγκαρ θα είναι παρόν και θα τοποθετηθεί. Έτσι λοιπόν τόσο τα κράτη-μέλη όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ε, ορίσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο. Με αυτό κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, εισαγάγει μέτρα παρεμβάσεως και σταθεροποίησης της αγοράς του χειρίου για να προστατευθούν οι γεωργικές, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προς συμφέρον ε, απάντων. Ωστόσο δεν μπορούμε και να λησμονούμε ότι θελήσαμε η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να προχωρήσει σταδιακά προς μεταρρυθμίσεις. Αυτό το επιδιώξαμε όλοι και υποστήριζε ανέκαθεν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ιδέα μιας αγοράς η οποία θα ε, λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις. Ε, βεβαίως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για ενίσχυση των συγκλήσεων, της συνοχής, αντιμετώπιση των κρίσεων, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι το συνεχές. άρνηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική λύση. Και εμεί θέλουμε μια πραγματική γεωργική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει σε επίγνωση των ε, ευθυνών τη και προσπαθεί να αναπτύξει μια κοινή γεωργική πολιτική μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο η οποία θα είναι ανθεκτική στις κρίσεις και μακροπρόθεσμα θα φέρει καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι είμαι στις παρατηρήσεις των βουλευτών που τοποθετήθηκαν σήμερα εδώ με τόσο περίφραστο τρόπο και βέβαια θέματα που έχουν να κάνουν και με την κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία και τις συνέπειες της κρίσης αυτής στον τομέα του χείριου κρέατος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε εξελίξεις. Ελπίζω ότι μπορώ να είμαι αισιόδοξο και να μην διαψευστώ στην αισιοδοξία μου αυτή. και άρα ε, μπορούμε να έχουμε σύντομα θετικές εξελίξεις και στον τομέα του χείριου κρέατος. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και έτσι ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης θα διατεθούν